δήλωση της Επιτροπής για το, για το σήμα προέλευσης. Το λόγο έχει η Επίτροπος Άστον. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχω τη δυνατότητα σήμερα να σας ε, απευθυνθώ στην Ολομέλεια παρουσιάζοντας έναν κανονισμό για το σήμα καταγωγής. Όπως μπορεί να ενθυμίσετε, γιατί το υποστηρίξατε, είναι μια πρόταση που χρονολογείται από το Δεκέμβριο του 2005 και που προέρχεται από το Σώμα των Επιτρόπων. Θυμούμε τη δήλωση της 6ης Ιουλίου του 2006 και την δήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου του 2007. Είχα το προνόμιο να συζητήσω αυτό το θέμα τον περασμένο μήνα στο Στρασβούργο με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μου τόνισαν ότι θα πρέπει να κινηθούμε ταχαίως για να εγκριθεί ο εν λόγω κανονισμός. Νομίζω ότι τα μέλη θα συμφωνούν ότι είναι θεμελιώδες η εμπορική πολιτική όχι μόνο να ενισχύσει τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η ελεύθερη αγορά αλλά να διευθετήσει και κάποιες ανησυχίες που γενεσιουργεί που γεννά η παγκοσμιοποίηση. Το σήμα καταγωγής αυτή τη φιλοδοξία έχει. Στη δήλωση ε, του 2003 τονίζεται το δικαίωμα των καταναλωτών να έχουν άμεση και σαφή πληροφόρηση για τις αγορές τους και περί αυτό ακριβώ πρόκειται ο κανονισμό αυτό. Ο στόχο έχει να δώσει στου Ευρωπαίου καταναλωτέ την ε, πλήρη εικόνα τη χώρα καταγωγή του προϊόντο που αγοράζουν. Γι' αυτό προτείνουμε υποχρεωτική ένδειξη τη χώρα καταγωγής ορισμένων εισαγόμενων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες και δεν τα καλύπτουμε όλα, καλύπτουμε αυτά που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον και αυτό μετά από ευρεία διαβούλευση με τον τομέα αλλά και τους πολίτες και τις ενώσεις καταναλωτών στο σεβασμό πάντα των κανόνων του ΠΟΕ και των αρχών που διέπουν ε, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Στη Ρωσία, στον Καναδά, στην Κίνα, στις ΗΠΑ υπάρχουν τέτοια μέτρα για τον εντοπισμό της καταγωγής του προϊόντος και ήδη ορισμένα προϊόντα που έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρουν αυτό το σήμα. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που θα υποχρεωθούν να, αποθέσουν σήμα καταγωγής δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο κόστος. Έχουν δε γίνει ε, πολλές συζητήσεις μέχρι τώρα στο Συμβούλιο για την πρόταση της Κομισιόν. Δεν έχουμε πείσει ακόμα όλα τα κράτη-μέλη που φοβούνται το διοικητικό άχθος και την οικονομική επιβάρυνση ότι ενδεχομένω αποδειχθεί μεγαλύτερα του ωφέλους. Εμείς έχουμε λάβει υπόψη μας όλες αυτές τις ανησυχίες και προσφάτως υποβάλαμε συγκεκριμένε προτάσεις για να υπερπηδηθούν αυτά τα προβλήματα και να διασκεδαστούν αυτές οι ανησυχίες. Δεν είναι νέα πρόταση, είναι μια απόπειρα εξέβρισης κοινού παρονομαστού και άρα ε, συμβιβασμού. Το ε, έγγραφο συζητήθηκε στην Επιτροπή 133 στις 23 Οκτωβρίου του 2009 Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη-μέλη να σκεφτούν το ενδεχόμενο μείωση των προϊόντων που καλύπτονται. Δηλαδή, μόνο προϊόντα της, που φτάνουν μέχρι τον τελικό καταναλωτή, στην τελική τους μορφή. Αλλά αποκλείονται. Η Κομισιόν τώρα όμως προτείνει να συμπληρωθούν μόνο τα αγαθά που μπορούν να βρουν έτοιμα σε καταστήματα λιανικής πωλήσεω ή καταναλωτή. Τώρα, έχουμε εξαγγείλει και ένα πολιτικό πρόγραμμα. Οποιοδήποτε συνέχιση θα αντικείμενο αξιολόγηση των συνεπειών του αντικτύπου της προτάσεως. Έτσι, θα κάνουμε μια αξιολόγηση αυτού του αντικτύπου και από πλευρά κόστου και από πλευρά τιμή των προϊόντων και μπορεί να έχουμε και κάποιε ενδείξει για το πώ μπορούμε να τροποποιήσουμε την κάλυψη των προϊόντων στα πλαίσια του κανονισμού και του πεδίου εφαρμογή του. Τα κράτη-μέλη, με χαρά μου μπορώ να πω, ότι διακίνεται ε, θετικά ή τέλο πάντων επέδειξαν ενδιαφέρον του εγγράφου αυτού. Βεβαίω δεν έχουν διασκεδαστεί όλε οι ανησυχίε. Ορισμένα κράτη-μέλη εμένουν επί τη αρχή του ε, ε, επί της διαφωνίας τους. Όμως θα συνεχίσουμε το έργο τις επόμενες εβδομάδες, το έργο προσέγγιση των μεν με τους δε και εξέβρεσης συμφωνίας ακόμα και στα πλαίσια της Επιτροπής 133 και ειλικρινά πιστεύω ότι θα ανοίξει έτσι ο δρόμος για μια οριστική συμβαστική λύση. Όπως θα ξέρετε το νέο άρθρο 207 της Συνθήκης της Λισαβόνας δίδει στο Κοινοβούλιο νέα περισσότερη εξούσια στον τομέα της εμπορικής πολιτικής και η τροποποίηση του κανονισμού μπορεί να είναι η πρώτη απτή απόδειξη αυτών των νέων σας αρμοδιοτήτων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα σας τηρώ ενήμερους ανα πάσα στιγμή και προσδοκώ στην επόμενη φορά που θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο από τώρα γιατί θα ξεπεράσουμε την 12η κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα με την υπηρεσία διερμηνίας. Γι' αυτό παρακαλώ τηρήστε τα χρονικά όρια. Για το ΕΛΚ για δύο λεπτά η κυρία Μουσκαρντίνη αξιότιμε Πρόεδρε και για μας είναι πρόβλημα η υπέρβαση του ωραρίου. Όχι μόνο για τους διερμηνείς, όχι για μας. Αλλά πάντω το θέμα είναι πολύ σημαντικό γιατί μας απασχολεί από το 2005. Όπως πολύ σωστά είπε η επίτροπο, είναι πολλά τα χρόνια από τότε που οι βασικοί μας εμπορικοί εταίροι και ανταγωνίστε έχουν ένα σήμα καταγωγή για τα προϊόντα που εισέρχονται στην επικράτειά τους. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την πρόταση κανονισμού του 2005 ευρεία συνένεση και συμφωνία των καταναλωτών και των ε, περισσότερων κατηγοριών της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών ε, μένουμε ακόμα αδρανείς παρά δε και το γεγονός ότι πολλά στο κοινοβούλιο έχει φραστεί υπέρ αυτής της αγούσης δηλαδή το σήμα καταγωγής που αποτελεί ένα δικαίωμα του καταναλωτού και του πολίτη και που αν δεν υπάρχει στρεβλώνει τους κανόνες ε, της ε, αγοράς. Για τις δύο αυτές κατηγορίες προϊόντων που αναφέρθηκαν στον κανονισμό έγινε μια προσπάθεια να γίνει ένα πραγματικό στάδιο, μελέτη αντικτύπου. Ζητούμε από την Επίτροπο η συμβαστική αυτή πρόταση να λάβει την συνένεση που έχει λάβει τη συνένεση ενός τουλάχιστον κομματιού των κρατών μελών να αξιολογηθεί περαιτέρω μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της συναπόφασης να μπορέσουμε να έχουμε στοιχεία και της πρότασης κανονισμού του 2005. Ποιες εγγύησεις, ποια ηχέγγυα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάτι τέτοιο. Και τέλος, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για όσα κάνατε με μεγάλη αποφασιστικότητα και δραστηριοποίηση. Θα ήθελα να σας ε, θυμίσω να σας παρακαλέσω μάλλον να μου επιβεβαιώσετε αυτό που στείλατε σε μια γραπτή σας απάντηση σε ερώτημά μου στις 5 Νοεμβρίου. Δηλαδή, λέτε, η Κομισιόν θα συνεχίσει να υποστηρίζει την υιοθέτηση της πρότασης υποκρισίας για το 2005 και θα συνεχίσει αποφασιστικά μάλιστα σε αυτή την οδό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Μουσκαρντίνη. Για τους σοσιαλιστές ο κύριος Σούστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν είναι πρόθεσή μου αυτήν την προκεχωρημένη ώρα να κάνω ιστορική αναδρομή όλων των λόγων που βρίσκονται στην βάση του επανειλημμένου αιτήματό μας ως Κοινοβουλίο. Εγώ και η κυρία Μουσκαρδίνη είμαστε οι δύο επιζήσαντες, ε, οι μόνοι δύο ε, μετά το 2005 που υποστηρίξαμε ε, την πρόταση Μάντελσον του τότε Επιτρόπου. Η πρωτοβουλία που λάβατε για μερική τροποποίηση του κανονισμού μπορεί να τύχει υποστηρίξεις και πρέπει και στην Επιτροπή 133 να γίνει δεκτή. Λυπούμεθα που στο βήμα αυτό στην Επιτροπή 133 δηλαδή πολλά κράτη-μέλη εξέφρασαν πάλι ανησυχίες και επιβεβαίωσαν την ε, άρνησή τους ε, όπως ε, η Βρετανική κυβέρνηση. Θέλουμε απλώς να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το αίτημα βασίζεται όχι σε προστατευτισμό. Δεν θέλουμε με τεχνητή αναπνοή να σώσουμε επιχειρήσεις που δεν είναι ανταγωνιστικές. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Θέλουμε να θέσουμε στην προσοχή όλων το θέμα της υγείας, του περιβάλλοντος και μιας πραγματικής αμοιβαιότητας της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό το οποίο λείπει σήμερα και δεν λείπει μόνο έναντι των πιο ευάλωτων υποκειμένων ή αντικειμένων του παγκοσμίου εμπορίου υπο, ε, ε, λείπει από όλου. Και από την Ινδία και από τη Βραζιλία και από, την, ε, από τους μεγάλες τέλος πάντων ανταγωνιστικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η κοινότητα έχει πρόβλημα να υπερασπίσει τα θεμητά της δικαιώματα. Εγώ θέλω το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει πλήρως τις πρωτοβουλίες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θελήσει να αναλάβει, όποιες και αν είναι και θέλουμε, θέλουμε οι δεσμεύσεις που ανέλαβε πριν από κάποιες εβδομάδες να φτάσουν μέχρι τέλους ακόμα και αν χρειαστεί, αν αποδειχτεί, να αναβληθεί η ολοκλήρωση της διαδικασία και να περιμένουμε τη θέση ισχύ της ε, ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Για τους Δημοκράτες και Φιλελεύθερους, για ένα λεπτό, ο κύριος Ρινάλντι. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, παρότι συμφωνώ με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες και με την κυρία Μουσκαρντίνη. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τον Ιταλο Καλβίνο που περιγράφει το Big Bang ως μια άμορφη μάζα που δεν ξέρουμε τίποτα για κανένα στοιχείο και την προέλευσή του. Αν θέλετε να το κάνετε έτσι, ε, είναι σαν να μην κάνετε διάκριση μεταξύ πίτσας και ταλιατέλων ή ταλιατελών τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τα χαρακτηριστικά από τα οποία αποτελούνται τα διάφορα προϊόντα. Εμείς ε, επιτιθέμεθα εναντί του συστήματος των ελεύθερων ανταλλαγών αλλά και της διαφάνειας και της ανιχνευσιμότητας των προϊόντων, της έλλειψης δηλαδή. Δεν είναι πρόβλημα διεθνούς εμπορίου όσο προστασία του καταναλωτού. Αυτό λέμε. Και υποστηρίζουμε την πρόταση του 2005 και επαναλαμβάνω, συμφωνώ με την Κριστιανά Μουσκαρδίνη και τα ερωτήματα που σας έθεσε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Ρινάλντι για τους πράσινους. Ο κύριος Καρλ Σλίτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επίτροπο για την ε, πρόταση αυτή. Νομίζω πως επιτέλους η Κομισιόν τόλμησε να αντιταχθεί στο Συμβούλιο και σας ευχαριστούμε. Διαπιστώνουμε πως δεν λειτουργεί μια αγορά εάν δεν έχουν πληροφορίες οι καταναλωτές για να λάβουν μια απόφαση. Είναι αναγκαίο να έχουμε αυτή τη σήμανση για την προέλευση. Δεν πρέπει να έχουμε εξαιρέσεις για τις χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνία ελευθέρου Να ισχύουν τα ίδια για όλους. Κόστος, το υψηλό κόστος σημαίνει πως ούτως ή άλλως πάρα πολλά προϊόντα σήμερα έχουν ε, σήμανση. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Το έχουμε δει αυτό και με άλλη σήμανση. Μας το έχουν πει και βλέπουμε πως δεν ήταν τόσο ακριβή τελικά. Κατά κανόνα δεν μιλάμε για προϊόντα τα οποία είναι πλαστά. και πάρα πολλά σημαντικά προϊόντα δεν δε συμπεριλαμβάνονται καν. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Σόλτς. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η ομάδα μου, η Γκουε, θεωρεί πως η σήμανση των προϊόντων προέρχονται εκτός της Ένωσης είναι κάτι το επίγον. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο και απορριθμισμένο κόσμο πρέπει να επιτρέψουμε στον καταναλωτή να ξέρει από πού προέρχεται ένα προϊόν και τι αγοράζει. Είναι λοιπόν ένα τομέα στον οποίο οι καταναλωτές καταλαβαίνουν τι εστί Ευρώπη και έτσι μπορεί να συνεισφέρει η Ευρώπη στο διεθνές εμπόριο. Συμφωνώ με τους συναδέλφους μου λοιπόν πως πρέπει να ακολουθήσουμε την υιοθέτηση του 2005. Και αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να αγγιηθούμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Για να βοηθήσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ευρώπης, καλούμε Κομισιόν και Συμβούλιο να υποβάλουν προτάσεις προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση στην πολιτική μας. Και εδώ το διεθνές εμπόριο μπορεί να συνεισφέρει στη διεθνή ειρήνη. Για δύο λεπτά η ναι. κυρία Κομή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς ε, Ανήκουμε σε ένα βιομηχανικό σύστημα όπου η φήμη των προϊόντων και το καλό του όνομα εξαρτάται πολύ από την ε, παραγωγική τους διαδικασία. Μπορούμε να δώσουμε χέγγια στους ε, καταναλωτές μας ότι ελέγχουμε τα προϊόντα μας που είναι υψηλή ποιότητα. Εάν θέλουμε αυτό να συμβαίνει και για τα εισαγόμενα προϊόντα, θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν πλήρη επίγνωση του τι παράγουμε, αλλά και το τι εισάγουμε και από πού το εισάγουμε. Για να επιτύχουμε το στόχο αυτό χρειαζόμαστε κάτι απλούστατο, μεν βασικότατον δε, τη διαφάνεια. Η αρχή της διαφανείας είναι στην βάση των κανόνων της ετικετοθεσίας και επισήμανσης καταγωγής που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο ήδη από το 2006 και που χρησιμοποιείται στις μεγαλύτερες αγορές ήδη όπως ανέφερε η Επιτρόπος από τη ΣΥΠΑ, το Μεξικό, την Κίνα. Παρ' όλα αυτά το Made in, το Made είναι δεν έχει ακόμα ευλογηθεί από πολλά κράτη-μέλη. Αν δεχόμαστε ανεξάρτητα από την ποιότητα του, την εισαγωγή των προϊόντων, ο καταναλωτής αν μη τι άλλο πρέπει να το ξέρει ότι αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε στην τάδε ή τη δίνα χώρα για να μπορέσει να επιλέγει εν πληρή επιγνώση. Η διαφάνεια δεν είναι υπερβολή δεν είναι προστατευτισμός. Δεν αυξάνει τις δαπάνες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν δεν υπάρχει ένδειξη καταγωγής για τα εισαγόμενα στην Ευρώπη προϊόντα, αντίθετα με αυτό που γίνεται στην Κίνα, τη ΣΥΠΑ και την Αυστραλία, θα καταστήσει πιο δύσκολη την κατάσταση από πλευρά ανταγωνισμού για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Για όλους αυτούς τους λόγους, ένα προϊόν που θα εφέρει αυτή τη σήμανση είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα προς την αναγνώριση όλων των προϊόντων σε επίπεδο κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ακόμη. Για δύο λεπτά ο κύριος Αρίφ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι η πρώτη συζήτηση που κάνουμε για την επισήμανση της προέλευσης, αλλά θα ήθελα να επιμείνω όπως και οι συνάδελφοι στην ανάγκη να υπάρξει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το Made In. Υπήρξε το ψήφισμα του συναδέλφου μας Μπαρόν Κρέσπο αλλά δεν εγκρίθηκε ο σχετικός κανονισμός στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα όχι μόνο για τον Ευρωπαίο καταναλωτή και την καταναλώτρια αλλά και για τις βιομηχανίες διότι η προέλευση ορισμένων προϊόντων από τρίτες χώρες είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζει ο καταναλωτής και η καταναλώτρια. Σε τομείς ευαίσθητους όπως η ένδυση ή τα δερμάτινα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο καταναλωτής την προέλευση του προϊόντος για να διατηρηθεί αν θέλουμε η βιοτεχνία στην Ευρώπη θα ήθελα να επιμείνω ότι πρέπει να επιδείξετε μεγαλύτερη φιλοδοξία κυρία Επίτροπε και να μην ικανοποιήσετε μόνο τα αιτήματα των χωρών μελών μειώνοντας την ποιότητα του προϊόντος ώστε να μπορούν να εισάγονται τα συστατικά του από αλλού και ε, μετά να θαμπάρετε made in Europe. Δεν επανέρχομαι λοιπόν σε αυτά που είχαμε πει στο παρελθόν για τη βελτίωση και απλοποίηση των κανόνων της ταύτισης της προέλευσης, αλλά ζητούμε ενίσχυση των δικτύων ελέγχου γύρω από τη Μεσόγειο. Κατά την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας θα έχουμε και εμείς περισσότερες δικαιοδοσίες και επομένως η Κομισιόν θα μπορεί να υπολογίζει, σας το βεβαιώνω κυρία Πρόεδρε, στη στήριξή μας αλλά και στον έλεγχο για την ποιότητα και προς του καταναλωτού και της καταναλωτρίας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ενά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνόδελφοι, το Made in δεν είναι απλώς θέμα σήμανσης, αλλά πρέπει να γίνει ολόκληρη έννοια και υπόδειγμα σεβασμού των κανόνων που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και μιας υπεύθυνη βιομηχανικής τάσης, οικονομικής τάσης. Γιατί αν μόνο μας κριτήριο είναι το κέρδος, τότε θα καταλήξουμε σε παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων συστηματικά. Τα πολυτελή προϊόντα τη χάνουν συνεχώς μιμήσεων και πάντοτε βάζουν το κέρδος ως πρώτο κριτήριο και από αυτά ζημιώνεται κυρίως ο καταναλωτής και η καταναλώτρια και οι θέσεις εργασίας. Με την ετικέτα Made in Europe θα μπορεί ο καταναλωτής και η καταναλώτρια να έχει την επιλογή να γνωρίζει ότι υπάρχει σεβασμός των κανόνων εργασίας και μιας υπεύθυνης διαχείρισης και πάνω απ' όλα να την χάνει του σεβασμού των θέσεων εργασίας. Ο κύριος Φέλνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, όσοι θέλουν προστατευτισμό δεν το ομολογούν και όλα σκρύβονται πίσω από άλλα πράγματα. Το σήμα της προέλευσης είναι ένα από αυτά. Τον Ιούνιο του 2006 εδώ στο κοινοβούλιο είχα ήδη μιλήσει για αυτή την πρόταση. Και τότε εξαφανίστηκε και πήγε στον κάλαθο των αχρήστων αυτή η πρόταση. Και ξαναγίνεται τώρα προσπάθεια ε, με αφορμή τη συμφωνία με την Κορέα να επανέλθει επιτάπητος. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι αξιοπρεπή πράγματα αυτά. Τόσα χρόνια ε, αφού του προσπαθήσαμε να σταματήσουμε αυτή την πρόταση. Έρχονται τώρα και μας λένε πως το ζητάνε οι καταναλωτές. Και να έχουμε διαβουλεύσεις. Ποιος το ζητάει. 86% των ετοιμάτων προέρχονται από την Ιταλία και μόνο. Και δεν μπορούμε να λέμε πως κάθε επιχείρηση πρέπει να το κάνει αυτό. Δεν χρειάζεται καν. Πρέπει να έχουμε τις ε, σχετικές πληροφορίες και ε, εδώ πέρα όμως δεν είναι ο στόχος καν ε, η προέλευση. Δεν προστατεύεται έτσι ο καταναλωτής. Ο δε άλλος μύθος είναι πως θα ενισχυθεί η δύναμη του Ευρωπαίου καταναλωτή ή οτιδήποτε άλλο. Ε, βλακίες. Μόνο οι ανοιχτέ αγορές οδηγούν σε ανταγωνισμό και η Ευρώπη δεν είναι ε, τίποτε άλλο. Είναι μια ανοιχτή αγορά. Δεν είναι ανάγκη τώρα να οδηγούμαστε σε προστατευτισμό. Πρέπει να έχουμε τους ίδιους κανόνες για όλους. Έχουμε ε, αυτή την πρόταση εδώ πέρα. Τώρα τι να πω. Εμείς θα πάμε κόντρα στον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ. Μινούτο. Για ένα λεπτό, η κυρία Μαγκίνες. ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ήδη σχετική σήμανση στα τρόφιμα και σε άλλα προϊόντα, δεν είναι τίποτα το καινούριο. Το πρόβλημα με κάποιες από τις ετικέτες στα τρόφιμα είναι πως δεν είναι ακριβής. Οπότε ό,τι κάνουμε εδώ πέρα σε αυτή την πρόταση, ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να μπορούμε να διαπιστώνουμε την αλήθεια αυτών που αναγράφονται στην ετικέτα και να έχουν τις πληροφορίες που ίσως να θένει οι καταναλωτές. Συγκεκριμένο ερώτημα τώρα. Εμένα μου τηλεφώνησε κάποιος ε, κατασκευαστής προϊόντων εντός της ε, Ένωσης και μου με ρώτησε εάν εξετάζουμε μια ετικέτα Made in European Union. Ίσως η Επίτροπος θα μπορούσε να μου απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Για ένα λεπτό ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό το επίμαχο ζήτημα. Καθώς μας απασχολεί πάρα πολύ στην Ιρλανδία και κάθε φορά που ακούμε τον επικεφαλής των αγροτών μας λέει πόσο δύσκολο είναι να έχουμε επαρκή σήμανση. Μπορούν να έρθουν προϊόντα στην Ιρλανδία, να τους βάλουν λίγο πιπέρι εκεί πέρα κάτι μπαχάρια και να είναι made in Ireland. Πρόκειται για εξαπάτηση του καταναλωτή. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν την χώρα προέλευσης και επεξεργασίας του προϊόντος. Και η πρακτική αυτή θα σταματήσει. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη σήμαση για να ξέρω καθένας από πού προέρχεται το προϊόν. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό. Ο κύριος Σιλβέστρης. Κυρία Επίτροπε, σαφήνεια, σαφήνεια, σαφήνεια. Αυτό ζητεί η αγορά σήμερα για κανόνες που να διασφαλίζουν τη διαφάνεια υπέρ του καταναλωτού. Η ελευθερία αγοράς δεν είναι ανεξέλεγκτη. Θα πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θα δώσουν το δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέγει εν πλήρη επιγνώση. Αυτό ζητούμε σήμερα. Στην κρατική τηλεόραση της χώρας μου πολλές φορές δημοσιεύονται έρευνες δημοσιογραφών και ε, δημοσιογράφων και ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα οποία πολλά προϊόντα χρησιμοποιούν τοξικές ουσίες ε, ε, με άθλες συνθήκες εργασίας, παιδική εργασία, ακόμα και σκλαβιά χρησιμοποιείται για να κατασκευαστούν πολλές φορές τέτοια προϊόντα. Θα τα δεχτούμε εμείς αυτά στην Ένωση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υποστηρίζω αποφασιστικότητα και επιγόντως την προσπάθεια υιοθέτηση κανόνων που θα δώσουν δυνατότητα στον καταναλωτή να μπορεί να επιλέγει το προϊόν που θέλει να αγοράσει εν πλήρη επιγνώση. Ευχαριστώ κύριε Σιλβέστρης, η κυρία Επίτροπος. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους όσους ε, συνέβαλαν στην σημαντική αυτή συζήτηση επί του σημαντικού αυτού θέματος. Να ξεκινήσω με αυτά που είπε η κυρία Μουσικαντίνη. Ότι τρενάρει αυτή η διαδικασία, ότι καθυστερεί. Εγώ, στη διάρκεια της θητείας μου ως Επιτρόπου, θέλησα πάντα να μιλώ με τα κράτη-μέλη για τα θέματα που τους ανησυχούν και να αντιδρώ όταν βλέπω κάτι σημαντικό. Αλλά η πραγματικότητα της πολιτικής ζωής είναι ότι εξαρτώμαι από το Συμβούλιο για να περάσω μία πρόταση. Όταν δεν υπάρχει σαφής πλειοψηφία στους κόλπους του Συμβουλίου, θα πρέπει να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω για να μην πάει χαμένη όλη αυτή η προσπάθεια. Και θεώρησα στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι έχουμε τη δυνατότητα, έτσι, επιφέροντας κάποιες ίσονος σημασίες αλλαγές να διασκεδάσω τις ανησυχίε των κρατών μελών και να ξαναπροσπαθήσω να λάβω το πράσινο φως. Ιδιαίτερα στο τέλος της θητείας αυτής της Επιτροπής <laughs> στη δική μου περίπτωση και πέραν του τέλους της θητείας αυτής της Επιτροπής. Δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ ότι θα επιτύχω, αλλά εξαρτώμαι δυστυχώς ή ευτυχώς από το Συμβούλιο. Πάντως έχω αναλάβει δέσμευση να συνεχίσω γιατί είμαι πραγματικά πεπισμένη είμαι πραγματικά πεπισμένη ότι το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολλά μέλη ανέφεραν συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τους καταναλωτές και την ευκαιρία που έχουμε εδώ για διαφάνεια και σαφήνεια να δώσουμε πληροφορίες σαφής και διαφανής στον καταναλωτή. Ελεύθερο εμπόριο όμως δεν σημαίνει μόνο ελευθερία, συμφωνώ, σημαίνει και διαφάνεια και ενημέρωση του καταναλωτού. Είναι έννοιες και αρχές που πάνε χέρι-χέρι. Συμφωνώ απολύτως και όσοι το είπαν νομίζω ότι άγγιξαν την καρδιά, τον πυρήνα της προσπάθειάς μας. Σε όλες τις χώρες γίνεται αυτή η προσπάθεια στις περισσότερες χώρες γνωρίζουν οι καταναλωτές από πού αγοράζουν κάτι. Και εγώ είμαι καταναλωτής. Και γνωρίζω ότι η σχέση του καταναλωτού με την αγορά περνάει και από αυτό. Έχουμε ευθύνη λοιπόν να επιφέρουμε αυτή τη διαφάνεια. Είναι πολύ σημαντικό. Και να μην τη φοβόμαστε. Γιατί αν τη φοβηθούμε κάποιο λάκκο έχει φάβα. Αν φοβόμαστε τη διαφάνεια, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Κύριε Σόλτς, για την επέκταση, επέκταση του καταλόγου των ε, προϊόντων που καλύπτονται. Κοιτάξτε, δεν είναι οριστικό ο κατάλογο. Εμεί προσπαθούμε απλώ να υπερβάλλουμε έναν ρεαλιστικό κατάλογο. Αλλά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το συζητήσουμε περαιτέρω. Τώρα, για το αν είμαστε ε, αρκετά φιλόδοξη. Κάποιο συνάδελφο, ο κ. Σαρίφ, είπε ότι θα πρέπει να νερώσουμε το κρασί μα. Όχι, δεν θέλω να νερώσω το κρασί μα, την πρότασή μα δηλαδή. Ρεαλιστή θέλω να είμαι. Και δεν θέλω κανείς αναπολώντας ή αξιολογώντας την κατάσταση να μου προσάψει ότι θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι που δεν έκανα. Μπορούμε όμως αυτά τα πιο λεπτομερή ζητήματα να τα ξανασυζητήσουμε στα πλαίσια του πιλωτικού αυτού προγράμματος για να δοκιμάσουμε, να τεστάρουμε την διαδικασία αυτή. Και τα θέματα EuroMed τα εξετάζουμε. Είναι κομμάτι της συζήτησης όπως ξέρετε και δέχομαι και αυτό που είπατε για την προστασία των ε, θέσεων απασχόλησης Ξέρετε ότι προστασία δεν σημαίνει προστατευτισμός, το έχω πει πολλάκις. Και δεν μπορεί το εμπόριο να τα αγνοεί όλα αυτά. Κύριε Βανέλη, είπατε ότι δεν φέρθηκα σωστά. Δεν νομίζω ότι λέγεται αυτό σε ένα ημικύκλιο. Πρέπει όμως να απαντήσω. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εγώ προσπαθώ να κάνω για όλες τις πτυχές της εμπορικής πολιτικής είναι να είμαι σε επαφή με όλους τους φορείς. μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ας πούμε, μας ανησυχεί πολύ ότι θα πρέπει να έχουν πραγματικές ευκαιρίες να ξεπεράσουν αυτό το 3% του μεριδίου αγοράς που έχουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην αφήσουμε κανέναν εκτός και να λύσουμε τα προβλήματα που δεν έχουμε επιλύσει μέχρι τώρα. Δεν είναι το μόνο θέμα βέβαια, αλλά θεώρησα ότι είναι μια ευκαιρία να το επαναφέρω στο προσκήνιο. Είναι θέμα ισότιμης ε, μεταχείρισης όλων, είναι θέμα ε, προστασίας των καταναλωτών, είναι θέμα διαφάνειας και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας αυτή να κάνουμε ακόμα πιο ε, οι συνενετικές προτάσεις. <clears throat> Τέλος, για το Made in European Union διαβουλευτήκαμε με τις επιχειρήσεις δεν προκρίθηκε η ιδέα αναφέρθηκε ότι θα ήταν δαπανηρή δεν την ε, ε, προέκρινε κανείς ευχαριστώ εγώ ευχαριστώ κυρία Επίτροπε έκλεισε αυτό το σημείο θα ψηφίσουμε στο ενεπόμενη ολομέλεια η, επόμενη ολομέλεια είναι αύριο στις 12 Νοεμβρίου 9 με 1. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί.